Καλησπέρα και καλώς ορίσατε στην κοινή συνεδρίαση αυτή με την ε, Επιτροπή Ανάπτυξης και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης είναι το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ε, αν δεν έχετε οποιαδήποτε ένσταση, είναι εγκριθεί η ημερήσια διάταξη ω έχει. Σας ευχαριστώ και να περάσουμε στο δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ανακοινώσεις του Προέδρου, δεν έχω ανακοινώσεις να κάνω. Και να συνεχίσουμε λοιπόν στο 3 της ημερησίας διάταξης και ο λόγος τον οποίο βρισκόμαστε όλοι εδώ σήμερα το απόγευμα, ανταλλαγή απόψεων με τον Αμπιταλά Χαντοκ, Πρωθυπουργό του Σουδάν. Συνάδελφοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους σας σε αυτή την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Εξωτερικής Ανάπτυξης για να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό του Σουδάν. Ξέρετε ότι έχουμε πολλά μέλη εδώ που παρακολουθούν το θέμα αυτό, παρόλο το γεγονός ότι έχουμε διακοπές και αργία σήμερα. Επίσης μεταδίδεται στο διαδίκτυο η σημερινή συνεδρίαση και έχουμε και διάφορους ε, βουλευτές μαζί μας. Ε, Πρωθυπουργέ, εξ ονόματος και των δύο επιτροπών, θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμότατα εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Η παρουσία σας εδώ πιστοποιεί τι σημαντικέ πολιτικέ αλλαγέ τι οποίε έχει περάσει τον τελευταίο, μήνε στο Σουδάν, ε, η κυβέρνησή σα ορκίστηκε και έτσι σηματοδότησε μια νέα εποχή στο Σουδάν και προσβλέπουμε να συζητήσουμε μαζί σα το μέλλον τη χώρα σα και τι σχέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Βιτχολτ Γιάν Βασκισκόφσκι που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροφής Εξωτερικών Υποθέσεων. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τόμπε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον κύριο Πρωθυπουργό του Σουδάν στη σημερινή συνεδρίαση των Επιτροπών μα. Η υπογραφή τη συνταγματική διακήρυξη τη 4 η Αυγούστου 2019 αποτελεί μια επιτυχία για το λαό του Σουδάν που επιθυμεί ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία. Και εμεί άλλωστε το ίδιο ευχόμαστε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Παρακολουθήστε, να, την μεταβατική αυτή περίοδο και υποστηρίζει τις προσπάθειες του Σουδάν για να πετύχει τη δημοκρατία. Η κυβέρνησή σας, τις οποίες και εγγύεστε, αποτελεί κλειδί για την επίτευξη του στόχου αυτού και για την δημιουργία κράτους δικαίου στη χώρα σας. Ο δρόμος λοιπόν δεν θα είναι εύκολος σε καμία περίπτωση. Είναι όμως κρίσιμη σημασία για το μέλλον της χώρας σας. Να συνεχιστούν λοιπόν αυτές οι ε, μεταβατικές ε, θεσμικέ ρυθμίσεις για να συνεχίσουν το έργο τους και να ακολουθούν τα καθήκοντά των. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε το Σουδάν και θα συνεχίσει να το κάνει προς όφελος του λαού του Σουδάν. Σας ευχαριστώ και τώρα θα ήθελα να ξαναδώσω το λίγο στον κύριο Τόμπε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαζευκόσκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατήρησε τη δεσμευσή της ε, για το λαό του Σουδάν παρά τις πολιτικές ε, ασυμφωνίες με την προηγούμενη κυβέρνηση και αποτελεί ένα από τους βασικούς δωρητές συνεργασία και ανθρωπιστικής βοήθειας στο Σουδάν. Από το 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει πάνω από 188 εκατομμύρια ευρώ στο ευρωπαϊκό καταπίστευμα για την Αφρική που θέλει να αντιμετωπίσει τις βασικές αιτίες αποσταθεροποίησης, εκτοπισμού και παράνομη μετανάστευση. Παρά τα προβλήματα που υπήρχαν σε ό,τι αφορά την ε, ανθρωπιστική πρόσβαση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παρέχει ανθρωπιστική αρρωγή ύψου 463 εκατομμυρίων ευρώ από το 2011, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επιστημιστική ασφάλεια, την ασφάλεια των τροφίμων. Οι πρόσφατε βελτιώσει ό,τι αφορά την πρόσβαση είναι κάτι το πολύ καλοδεχούμενο. Η ανθρωπιστική κατάσταση εξακολουθεί να είναι ε, τραγική σε διάφορε περιοχέ τη χώρα σα, με εκατομμύρια πρόσφυγε και ιστορικά εκτοπισμένου. Ανυπομονούμε να συζητήσουμε μαζί σα για το πώ θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αυξήσει την ανθρωπιστική τη δράση στο Σουδάν. Άλλα θέματα κοινού συμφέροντο, το οποίο θα μπορούσαν να βελτιωθούν από στάντορη συνεργασία μεταξύ ημών και ημών, είναι η συνεργασία και η ανάπτυξη, η περιφερειακή ενσωμάτωση, Ολοκλήρωση, το εμπόριο, η καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο, η ασφάλεια και η μετανάστευση. Πρωθυπουργέ, αν υπομονούμε να ακούσουμε πώ εκτιμάτε εσεί την κατάσταση στη χώρα σα και να ακούσουμε τι δικέ σα απόψει για τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Σουδάν. Έχετε το λόγο, κύριε Πρωθυπουργέ. Thank uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλου, Καλό βράδυ. αξιότιμα μέλη και των δύο επιτροπών ανάπτυξης και εξωτερικών σχέσεων ε, είναι τιμή για μένα και χαρά που έχω την ευκαιρία να σας επευθύνω το λόγο εκ μέρους του Συμβουλίου Κυριαρχίας του Σουδάν να εκφράσω πρώτα απ' όλα την ευγνωμοσύνη μας και τις ευχαριστίες μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την συνεχιζόμενη υποστήριξή της στον αγώνα του Σουδανικού λαού κατά τη διάρκεια της ε, δικτατορίας. Επίσης μας είχατε υποστηρίξει και αυτό μας επέτρεψε να φτάσουμε στη φάση που βρισκόμαστε σήμερα. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά και σας βεβαιώ ότι εκτιμά ιδιαίτερα ο Σουδανικός λαός την υποστήριξη αυτή. Ήθελα σε αυτή τη σύντομη εισήγηση να σας ε, διαβιβάσω τις προκλήσεις και τις προθέσεις μας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και τις προσδοκίες που έχουμε από τη σχέση αυτή. Επιτρέψτε μου λοιπόν πολύ σύντομα να ε, περιγράψω τις προτεραιότητες, αλλά πριν από αυτό να σας πω πώς βλέπουμε τις εξελίξεις των, τελε... των τελευταίων 7-8 μηνών στο Σουδάν Είμαι βέβαιος ότι έχετε παρακολουθήσει τι συνέβη. Οι αλλαγές είναι πραγματικά ευρύτατες και αφορούν στο σύνολο της χώρας. Στην πρόσφατη ιστορία μας τα τελευταία 60 χρόνια, είχαμε πάρα πολλές μεταβατικές φάσεις στην περιοχή μας είχαμε ηγηθεί από το 64 στην προσπάθεια ανατροπής των δικτατοριών το 85 επίσης και αυτή τη φορά τελευταία το 19 στις προηγούμενες δύο ε, μεταπολιτεύσεις ε, είχε κυρίως εστιαστεί το φαινόμενο στην πρωτεύουσα ενώ τώρα είχαμε διαδηλώσεις εντυπωσιακότατες από το δυτικό Νταρφούρ στο βορρά, στην Ανατολή, στο κέντρο, σε όλη τη χώρα και όλοι αυτοί κινήθηκαν προς την πρωτεύουσα. και είχαμε και ιδιαίτερότητε Έχουμε κρίση στην ευρύτερη περιοχή βέβαια, όπως γνωρίζετε, στη Λιβύη, στην Κεντρική Αφρική, στην Ιεμένη, στη Συρία, στη Σομαλία, μόνο αυτές έτσι αναφέρω. Η δική μας αλλαγή έγινε με ειρηνικό τρόπο και αντισταθήκαμε στο να αντιδράσουμε στις προκλήσεις του, της προηγούμενης κυβέρνησης. Επίσης ηγήθηκαν της προσπάθειας αυτής και της διαδήλωσης αυτής οι νεαροί και οι γυναίκες που ηγούνται όλες αυτής τις προσπάθειες. Ο λαός υπήρξε ιδιαίτερα ανθεκτικός όποτε ανησυχούσαμε ότι το κίνημα πήγαινε να σβήσει μας εξέπληξε με την ανθεκτικότητά του, με την επιμονή του και με τη συμμετοχή του συνόλου του πληθυσμού. Τώρα, οι προτεραιότητες αυτής της μεταβατικής φάσης, μετά από μακρά διαδικασία, έχουμε ε, φτάσει στο σημείο να έχουμε κάποιες ε, μεταβατικές διευθετήσεις με το Συμβούλιο της ε, κυριαρχία το Υπουργικό Συμβούλιο και την ηγεσία του δικαστικού σώματος. Η μεταβατική αυτή φάση ήταν στο πλαίσιο ελευθερία, ειρήνη και δικαιοσύνη που ήταν το βασικό μήνυμα του αγώνα μας αυτού. Με 10 προτεραιότητες λοιπόν, υπαριθμόν ένα, να σταματήσουμε τον πόλεμο και να οικοδομήσουμε μια βιώσιμη ειρήνη. Από την πρώτη μέρα ξεκινήσαμε την προσπάθεια αυτή και δεν ήταν κατά τύχη που η πρώτη μου επίσκεψη εκτός του χαρτού μου ήταν στην Τζούμπα, στο νότιο Σουδάν, θεωρούμε ότι είμαστε ένα έθνος σε δύο κράτη. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τον Νότιο Σουδάν. Και μας υποδέχθηκαν πολύ θερμά οι Νότιοι Σουδανοί με πολύ υψηλά ποσοστά που ψήφισαν υπέρ της ανεξαρτησίας αλλά έχουμε άνω των 2.000 χιλιόμετρων, 2000 χιλιόμετρων χερσαία σύνορα κοινή παράδοση, κοινή ιστορία αλλά και η επίσκεψη στη Τζούμπα ήταν μια ευκαιρία να ε, γνωρίσουμε και την ηγεσία των ένοπλων ομάδων που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο. Και μιλώντας μαζί τους, δεν είναι σαν να μιλάμε με κάποιον άλλον παρά με τον ίδιο μας τον εαυτό. Και στην συζήτηση μαζί τους είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να πετύχουμε γρήγορα ειρήνη, προσπαθώντας να επιλύσουμε προβλήματα ανθρωπιστικά, πρόσβασης, με διάφορες οδηγίες και διατάξεις για ομαλή πρόσβαση διασυνοριακά, για να επιτρέψουμε στην ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει εκεί που χρειάζεται. Ξεκινήσαμε επίσης κάποια, να αναλαμβάνουμε κάποια πρακτικά βήματα. Την περασμένη εβδομάδα ήμουν στον Ταρφούρ, στο El Fasher, και επισκέφθηκα τα κέντρα IDP. των εσωτερικά εκτοπισμένων πληθυσμών λοιπόν για να συνομιλήσουμε με τους επικεφαλείς των κέντρων αυτών η εντύπωση που είχα είναι ότι μπορούμε να επιτύχουμε την ειρήνευση και νομίζω ότι είναι μοναδική ευκαιρία για μας να το πετύχουμε αυτό. Επίσης, η δεύτερη προτεραιότητα είναι να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση και να αναβιώσουμε την οικονομία. Εδώ και 30 χρόνια τουλάχιστον αντιμετωπίζουμε κακοδιαχείριση, πολύ σημαντικές κρίσεις που εκφράζονται με εξαιρετικά υψηλές τιμές, εξαιρετικά υψηλό πληθωρισμό νομισματική κρίση, ο τραπεζικός τομέας σχεδόν έχει καταρρεύσει και επομένως προτεραιότητά μας είναι να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση, να αντισταθεροποιήσουμε και να θέσουμε τη χώρα σε μια κατεύθυνση ομαλοποίηση της οικονομίας γιατί το Σουδάν είναι πλούσια χώρα εφόσον διαχειριστούμε σωστά τους πόρους μας θα έχουμε το πλεόνασμα που θα μας χρειαστεί ώστε να το διοχετεύσουμε προς την ανάπτυξη, την οικονομική μεγέθυνση. Τρίτον, πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τους κρατικούς ε, θεσμούς. Και εδώ παραλάβαμε κατεστραμμένους, ε, υποβαθμισμένους θεσμούς. Τέταρτον, πρέπει να οικοδομήσουμε θεμέλια για την ομαλή λειτουργία του κράτους δικαίου, της διαφάνειας της δικαιοσύνης. Και ιδιαίτερα της δικαιοσύνης αυτής της μεταβατικής περίοδου, δηλαδή να έχουμε μια διαδικασία που θα μας επιτρέψει να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε να ικανοποιηθούν οι πολίτες που έχουν πληγεί, τα θύματα, ότι έχει υπάρξει δικαιοσύνη. Πέμπτον, να καταπολεμήσουμε τη διαφορά και να ανακτήσουμε κλεμμένα, κλεμμένη περιουσία. Δισεκατομμύρια δολάρια έχουν βγει από τη χώρα και τα έχουν κρύψει. Θα θέλαμε να τα, να τα ανακτήσουμε ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, επίγουσες οικονομικές μας και άλλες ανάγκες. Έκτον, θέλουμε να δουλέψουμε προς μία δίκαιη γυναικεία εκπροσώπηση, εκπροσώπηση των γυναικών στις κρατικές μας δομές, του θεσμούς. Και εδώ, στο Συμβούλιο Κυριαρχίας, που έχει 11 μέλη, ήθελα να σας πω ότι έχουμε δύο γυναίκες, μία εκ των οποίων είναι από την μειονότητα των κοπτών. Ε, και θεωρήσαμε ότι αυτό το θέμα θα ήταν ένας καλός τρόπος να αντιμετωπίσουμε και τα θέματα της διαφορετικότητάς μας. Ε, έχουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο τέσσερις γυναίκες. Η συνάδελφος εδώ είναι υπουργό ε, Κοινωνικής Ανάπτυξης. Επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά νομίζω για πρώτη φορά στην ιστορία μας έχουμε έναν επικεφαλής του δικαστικού σώματος που είναι γυναίκα. Προσπαθούμε να πληρώσουμε το νομικό συμβούλιο με τουλάχιστον 40% από τις θέσεις να, είναι, να πάνε σε γυναίκες. Νομίζω ότι είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν μας ικανοποιούν απολύτως, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε και άλλα θέματα για την εκπροσώπηση των νέων και των γυναικών. Για πρώτη φορά δώσαμε θέσεις αντιπριτάνεων στα πανεπιστήμια, σε γυναίκες και βλέπουμε την επίπτωση στις γυναίκες που πηγαίνουν, στα νεαρά κορίτσια που πηγαίνουν στα πανεπιστήμια. Και είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιες θέσεις σε γυναίκες στη χώρα μας. Πολλοί θα έλεγαν ότι αυτό είναι ένα εποχιακό φαινόμενο, αλλά μπορούμε να το υποστηρίξουμε βιώσιμα με την κοινή προσπάθειά μας για τα θέματα αυτά εκπροσώπησης. 8. Προσπαθούμε να έχουμε μια εξωτερική πολιτική ισορροπημένη χωρίς να παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά άλλων αλλά το καθεστώς για πάρα πολλά χρόνια κατέστρεψε τις εξωτερικές μας σχέσεις, αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Επίσης πρέπει να καλύψουμε το θέμα της ενεργείας για τους νέους. Πρέπει να δημιουργήσουμε ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, ένα περιβάλλον εντός του οποίου θα ξανακερδίσουν το μέλλον της χώρας ή οι νέοι μας και θα επιστρέψουν ίσως αρκετοί από αυτούς στη χώρα. Αντί να πηγαίνουν σε <clears throat> επικίνδυνες μεταναστεύσεις. Γιατί η φυγή των νέων μας είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα για μας. Και νομίζουμε με, μια σωστή συνεργασία μαζί σας μπορούμε <clears throat> να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη πολλών από αυτούς και να επιστρέψουν. Επίσης, προτεραιότητα μας είναι τα κοινωνικά θέματα Τα θέματα επίσης υγείας, παιδεία και καλύτερης διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων. Το καθεστώ χρησιμοποιούσε 70 με 80% των πόρων μας στα θέματα ασφαλείας. Η ειρήνευση θα μας επιτρέψει να αλλάξουμε την κατάσταση αυτή και να διοχετεύσουμε, να χρησιμοποιήσουμε μάλλον τους πόρους μας, να τους αναπτύξουμε προς πιο ωφέλιμε προσπάθειες, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη χωρίς καλύτερη χρησιμοποίηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Και τελευταία προτεραιότητα, θέλουμε να έχουμε μια συνταγματική διάσκεψη για να καλύψουμε προβλήματα διακυβέρνησης, εθνικής ταυτότητα, ανάπτυξης και να διοργανώσουμε εκλογέ που θα δώσουν την ευκαιρία στους πολίτες μας να εκφράσουν τη βούλησή τους να επιλέξουν την κυβέρνηση που επιθυμούν. Πρόεδρε, θα ήθελα τώρα να στραφώ στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, γιατί δεν θέλω να είναι υπερβολικά ρόδινη η εικόνα που σας περιγράφω. Δεν θα έλεγα ποτέ ότι τα ελέγχουμε όλα μετά την ανατροπή του δικτάτορα. Ε, το πρώτο που θέλω να πω είναι η πρώτη και μεγαλύτερη πρόκληση είναι να επιτύχουμε ειρήνη. Έχουμε πολλές ένοπλες ε, δυνάμεις, πάρα πολλούς ε, παράγονες παίκτες που διερματίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Έχουμε πολλές προκλήσεις, αλλά το βασικότερο είναι να επιτύχουμε την ειρήνη. Οι προκλήσεις και τα προβλήματα παραμένουν σημαντικά. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Κλίντον ήταν τότε, πριν από κάποια χρόνια, που κατά τη διάρκεια των, της προεκλογικής εκστρατείας είπε ότι το σημαντικότερο από όλα είναι η οικονομία. Η οικονομία παίζει ρόλο και αυτό ισχύει γιατί σε εμά σίγουρα παίζει ρόλο το θέμα του χρέους ε, και πάρα πολλά άλλα στην αφή. Αυτό που ενδιαφέρει κυρίως ε, είναι η οικονομία κατά τη διάρκεια της ε, μεταβατικής περίοδου. Οι κρατικοί θεσμοί είτε στον λοιπόν τομέα είτε σε θέματα ασφάλειας, εκεί υπάρχουν πολλά προβλήματα και είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείτε και τον κατάλογο των κρατών που χρηματοδοτούν ε, τους τρομοκράτες. Είναι ένας κατάλογος ε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς βρισκόμαστε σε αυτό τον κατάλογο, αλλά είναι πολύ σημαντικό για μας να βγούμε από αυτό τον κατάλογο και έτσι θα λυθούν πολλά ε, προβλήματα. Κατά το παρελθόν, ίσως να μπορούμε να καταλάβουμε γιατί μπήκαμε σε αυτό τον κατάλογο, αλλά σήμερα όμως πλέον δεν είμαστε χώρα που να στηρίζει τους ε, τρομοκράτες, καμία σχέση. Εμείς είμαστε μια χώρα που αγαπά την ειρήνη και πιστεύω ότι με τη δική σας την υποστήριξη θα μπορέσουμε να πείσουμε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αφαιρέσει το Σουδάν από αυτό τον κατάλογο. Συνεργαζόμαστε μαζί τους για το θέμα και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα που θα μας επιτρέψει και το να έλθουν επενδύσεις στη χώρα μας. Ε, το πρόβλημα βεβαίως είναι ότι έχουμε πάρα πολλές ε, ε, και υψηπετείς ε, προσδοκίες. Το να τις αντιμετωπίσουμε δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι είμαστε διαφανείς, ανοιχτοί και έχουμε και την υποστήριξη του λαού. Δεν θέλουμε να τους απογοητεύσουμε. Υπάρχει βέβαια κληρονομιά πολλών ετών, αλλά νομίζω ότι από κοινού θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Το θέμα το να μην υπάρχουν υποκλεισμοί, να υπάρχει ανταπροσωπευτικότητα, να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο για τη χώρα, αλλά να μπουν και τα θεμέλια για τη μετάβαση στη δημοκρατία. Και τώρα θα αναφερθώ στο τελευταίο κομμάτι των σύντομων παρατηρήσεών μου. Έχουμε προσδοκίες από πλευράς εταίρων μας και όπως είπα προηγουμένως κατανοούμε πολύ καλά την ε, συνεχή υποστήριξή σας ε, στην αντιμετώπιση των ε, προβλημάτων μας. Έχετε δει και εσείς κάποια δείγματα από τη δική μας την πλευρά. Νομίζω λοιπόν ότι από κοινού θα έχουμε μια καλύτερη στρατηγική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορέσουμε να μοχλεύσουμε πόρους, να αναζητήσουμε την ειρήνη. Σύντομα όμως, επιτρέψτε μου ε, να σας πω τι περιμένουμε εμείς από εσάς. Περιμένουμε την υποστήριξή σας στις ε, ειρηνευτικές ε, διαδικασίες, στις συζητήσεις μας. Περιμένουμε να στηρίξετε τη διαδικασία ειρήνης και να χρηματοδοτήσετε την ανάπτυξη μετά την επίλυση των συγκρούσεων. Να κινητοποιηθούν ανθρωπιστικοί πόροι προς ε, την κατεύθυνση του Σουδάν και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα το πρωί άκουσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν υποσχέσεις ε, να μας στηρίξουν με επιπλέον κονδύλια. Θέλουμε επίσης να μας βοηθήσετε για να αφαιρεθεί ε, το Σουδάν από τον κατάλογο κρατών που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία. Και μέσω, μακρο, μέσω μακροπρόθεσμα θέλουμε να στηρίξετε την οικονομία του Σουδάν μέσα από επενδύσεις, οικονομικές συνεργασίες, γιατί για μεγάλο χρονικό διάστημα η χώρα ήταν ε, αποκλεισμένη από ξένες επενδύσεις λόγω των πολιτικών που ακολούθησε το προηγούμενο ε, καθεστώς. Θέλουμε ευρωπαϊκό κεφάλαιο, επιχειρήσεις να επανέλθουν σε εμά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Μπορούν να κατασκευαστούν δρόμοι, λιμάνια, για υποδομές ε, ε, στον τομέα των ορυχείων, ε, στις, στα κοιτάζοντα πετρελαίου. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες στο Σουδάν. Επίσης, ελπίζουμε να μας υποστηρίξετε στην εξέλιξη και ανάπτυξη των ικανοτήτων μας, όπως είπα και προηγουμένως. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι το Σουδάν ε, προσβλέπει στην πλήρη συνεργασία με την διεθνή κοινότητα, με τους εταίρους μας και κυρίως ε, προσβλέπουμε στο να σφυριλατηθεί μια στρατηγική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να συνεργαστούμε για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα που προανέφερα. Αλλά το να ε, βοηθήσω στο Σουδάν σημαίνει ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα από κοινού, κάτω από στρατηγική σκοπιά, γιατί αυτό θα λύσει και πολλά άλλα προβλήματα. Ε, αν δεν ε, βοηθηθεί το Σουδάν, μπορεί να ε, μετακυληθεί αυτός ο σπόρος των συγκρούσεων σε γειτονικέ χώρες και αυτό θα ήταν πολύ άσχημο για όλη την περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ που μου δώσετε τη δυνατότητα να σας απευθύνω το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ για την εισαγωγή αυτή η οποία α, περιέχει πολλές προκλήσεις αλλά προφανώς και δίνει ελπίδα όμως. Να ξεκινήσει λοιπόν τώρα ο γύρος ερωταπαντήσεων, να ακούσουμε τους συντονιστέ, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα μέλη της Εξωτερικής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για να κάνουν ερωτήσεις και μετά το λόγο θα έχει και ο Πρωθυπουργός προφανώς. Οι συντονιστές. Ο κ. Γκάλερ, καταρχάς, από το ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ πολύ και καλώς ορίσατε κύριε Πρωθυπουργέ στο κοινοβούλιο μας. Χαιρόμαστε που έχουμε τη νέα κυβέρνηση του Σουδάν εδώ. Είμαι εδώ στο κοινοβούλιο 20 και πλέον έτη. Σε ό,τι αφορά και τις σχέσεις με την συγχωρησακή. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε μάλλον ε, πόσο συχνά έχουμε συζητήσει το θέμα του Σουδάν. Είχαμε συνομιλίες και με εκπροσώπους της χώρας σας τότε, εκπροσώπους της χώρας σας και ε, με άλλες αφρικανικές χώρες. Ήταν ευχάριστη η ανταλλαγή απόψεων. Είναι ευχάριστο το γεγονός που υπάρχει καινούριο και καινούριος αέρας και ελπίζουμε αυτό να διέπει και τις ε, σχέσεις μας. Ε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον προφανώς, αλλά όλοι μπορούμε να εργαστούμε για ένα καλύτερο μέλλον. Έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά θα πρέπει να περιοριστώ γιατί θα έχουμε και άλλους συναδέλφους που θέλουν να πάρουν το λόγο, αναφερθήκατε στον Ταρφούρ. Αυτό μας έχει απασχολήσει εδώ και χρόνια. Αναρωτιέμαι. Καταρχάς, τι συγκεκριμένα βήματα γίνονται σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τις διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις και με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναβαθμιστεί η κατάσταση εκεί. Αναφερθήκατε στους εσωτερικά εκτοπισμένους. Υπάρχει κάποιο σχέδιο να επανακατασταθούν κάπου. Τι μέτρα πέρα από τις επισκέψεις εκεί θα αναλάβετε για να δημιουργήσετε και πάλι ένα καθεστώς εμπιστοσύνης προς την κεντρική κυβέρνηση. Ένα άλλο θέμα στο οποίο ήθελα να αναφερθώ. Έχει να κάνει με τη σχέση σας με το Νότιο Σουδάν. Και δεν θα αναφερθώ στα γεγονότα εκεί, αλλά αυτό που είναι σημαντικό και για σας και για το Νότιο Σουδάν είναι η εξαγωγή πετρελαίου. Το πετρέλαιο είναι κυρίως ε, στο Νότιο, αλλά οι αγωγοί περνούν ε, από εσάς. Ελπίζαμε ότι σε κάποιο σημείο αυτό το αμοιβαίο όφελος ε, θα αναγνωριζόταν και από τις δύο πλευρές. Ε. Πού βρισκόμαστε στην παρούσα φάση. Προχωράνε οι εξαγωγές πετρελαίου. Υπάρχει κατανομή των κερδών. Λειτουργεί το σύστημα και για τις δύο πλευρές. Θα περιοριστώ σε αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χόλμαν δεν είναι εδώ, βλέπω. Αποχώρησε. Μάλιστα. Από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες ο κύριος Μίξερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρωθυπουργέ που μας το χρόνο για να μας ενημερώσετε για τις εξελίξεις στη χώρα σας. Προφανώς σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας Δύο ερωτήσει. Αναφερθήκατε εν συντομία στα δημοσιονομικά στη χώρα σας. Και προφανώς υπάρχει και το χρέος, υπάρχει και η περιορισμένη ικανότητα εισπραξης φόρου που προφανώς και εμποδίζει την κυβέρνηση να παρέχει τις απαραίτητες ε, υπηρεσίες που χρειάζεται να προσφέρει προς το κοινό. Αυτό αποτελεί και μεγάλη προσδοκία του κόσμου. Μπορείτε να μα πείτε σύντομα τι πρέπει να γίνει για να ρυθμιστεί αυτό το σκέλος. Δεύτερη ερώτηση από έναν εντελώς διαφορετικό τομέα. Εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες για μακρά χρονική περίοδο για τις διαφωνίες σε ό,τι αφορά τα ύδατα του Νείλου και το πώς θα κατανεμηθούν αυτά τα ύδατα. Υπάρχουν κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά το, α, τα αποθέματα. Θα ήθελα να ακούσω την ε, δική σας τοποθέτηση. Πώς μπορεί να επιληθεί αυτή η διαφωνία προκειμένου να μην προκληθεί καμία τριβή μεταξύ των τριών χωρών, αλλά για να προωθηθεί και η οικονομική ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Από τους Ελληνικούς και Δημοκράτες, ο κ. Σιγμαθαδίτης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, ως πρώην Πρωθυπουργός της δικής μου χώρας, της Πολωνίας, δεν μπορώ παρά να φανταστώ απλώς ε, τις τεράστιες δυσκολίες και την ευθύνη που βαρύνει τους ώμους σας. Ε, παρακολούθησα τις εξελίξεις στη χώρα σας, τις παρακολουθώ 40 χρόνια τώρα. Και είχα και προσωπικούς λόγους πριν από 40 χρόνια ε, στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας είχα την τιμή να έχω ένα φίλο, τον ε, κύριο Αμπτελ Μαλί Καλμπερέη από το Σουδάν που εκεί ε, έκανε το διδακτορικό του. Και από τότε είχα ένα προσωπικό ενδιαφέρον στην παρακολούθηση των εξελίξεων στη χώρα σας. Και έτσι είδα τα τελευταία 20 χρόνια τις δικτατορίες και τις ε, πολιτικές εξελίξεις. Άκουσα προσεκτικά τις προτεραιότητες που μας περιγράψατε για την ειρήνευση και την οικονομική ανάπτυξη ώστε να αντιμετωπίσετε τις βασικότατες προσδοκίες που έχουν από εσάς οι πολίτες και είναι πολύ σημαντικό. Στο δέκατο σημείο σας αναφερθήκατε στη δημοκρατία. Κατανοώ πόσο δύσκολο είναι κανείς να οικοδομήσει τη δημοκρατία με τέτοιες τραυματικές και τραγικές θα έλεγα εμπειρίες. Αλλά έχω δίκιο θεωρώντας ότι αυτές οι μαζικότατες διαδηλώσεις που κατέληξαν στην ε, κατάργηση, στην αποχώρηση του καθεστώτος δεν ήταν μόνο κατά Τη ίδια τη δικτατορία, αλλά και υπέρ του αιτήματο του λαού να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους, οι ελευθερίε τους και να οικοδομηθεί ένα δημοκρατικό σύστημα στη χώρα. Επίση, μπορείτε να μα πείτε σε ποιο βαθμό η εμπειρία της γειτονική σας χώρας, της Αιθιοπίας, θα μπορούσε να είναι ίσως ένα παράδειγμα. Γιατί η Αιθιοπία και το Σουδάν έχουν, ε, μοιράζονται μια πολύ δύσκολη ιστορία και ε, ε, γνώρισαν αρκετή επιτυχία στην μεταρρύθμιση του δικού τους πολιτικού συστήματος και ειρήνευσης με έναν από τους γείτονες. Εσείς θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να ακολουθήσετε αυτό το παράδειγμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ λέει ο Πρόεδρος. Θα ακούσουμε δύο ακόμα μέλη όπως και την Επιτροπή και την ΙΕΔ. Η κυρία Καμκούν είναι εδώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά κύριε Πρωθυπουργέ. Θα σας κάνω ένα δύσκολο ερώτημα. Και φαντάζομαι ότι θα σας είναι δύσκολο, γιατί όλοι ελπίζουμε να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, να ήταν διαφορετική η ιστορία και ίσως θα αισθανθείτε περίεργα, αλλά δεν πρέπει να λυπόμαστε για το μέλλον πολλών γυναικών και κοριτσιών στον κόσμο και στη δική σας χώρα, που είναι και η χώρα από την οποία προέρχομαι είναι η ένατη χώρα στον κόσμο ε, στον γάμο των ανηλίκων κοριτσιών. Μεταξύ των πρωταθλητών λοιπόν τους παιδικούς γάμους, στους γάμους με παιδιά. Ε, διάβασα πέρυσι ότι ε, στο facebook ε, είχαν στην ουσία πουλήσει ένα μικρό κορίτσι για να παντρευτεί. ή είχαν ανταλλάξει με 500 αγελάδες 10.000 δολάρια ώστε να γίνει η δέκατη σύζυγος κάποιου. Αυτό το μικρό κορίτσι. Και φέτος διάβασα ότι καταδικάστηκε σε θάνατο ένα κορίτσι ώστε να γιατί δολοφόνησε τον σύζυγό του ο οποίος την κακοποιούσε. Όλα αυτά σημαίνουν ότι ε, στη χώρα σας ε, δύο από τρεις χώρες χοντρικά έχουν αυτές τις ίδιες ευκαιρίες που είχαν και στον παρελθόν. Εγώ πιστεύω ότι όλες οι γυναίκες πρέπει να αισθάνονται προστατευμένες και ότι έχουν ίσα δικαιώματα. Και αυτό είναι ο μόνος τρόπος να κινηθείτε προς τα εμπρός στην έκφραση του Προέδρου Κλίντον «The economy stupid» πρέπει να προσθέσουμε και την υπενθύμηση για την κατάσταση των γυναικών. Πρέπει να έχουν ευκαιρίες να παρακολουθούν σχολικές και πανεπιστημιακές σπουδές και σας ρωτώ τι βήματα θα αναλάβετε ώστε να προστατεύσετε τα κορίτσια και τις γυναίκες σε ε, καταναγκαστικούς γάμους, πώς το νομικό σύστημα της χώρας σας θα προσαρμοστεί για να παράσχει την προστασία αυτή στις γυναίκες και στα ανήλικα κορίτσια. Πώς θα συνεργαστεί η κυβέρνηση του Σουδάν με τη UNICEF ή άλλους διεθνείς φορείς και με θρησκευτικές οργανώσεις ώστε να δώσει τις ευκαιρίες που αξίζουν στα κορίτσια, στις νέες γυναίκες. Μία στις δύο γυναίκες στην Μπουρκίνα Φάσο ε, υφίστανται αυτή τη μοίρα και θα την είχα υποστεί κι εγώ, αλλά εμένα ευτυχώ οι γονεί μου έστειλαν στο σχολείο. Πώ φαντάζεστε το μέλλον των γυναικών, των κοριτσιών στη χώρα σα, Γιατί χρειάζεται να συμμετάσχουν. Και επίση, πώ μπορούμε σε αυτό να σα βοηθήσουμε. Ε, ο πρόεδρος λέει, ο κύριος Μάντελ από το ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Με χαρά σα έχουμε εδώ μαζί μα κύριε Ποθεπουργέ. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να συζητήσουμε, να μιλήσουμε και να κοιτάξουμε προς την ίδια κατεύθυνση και ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τη σχέση σας με Ρωσία και Κίνα. Θα ήσασταν σε θέση να μας δώσετε κάποιες σκέψεις σχετικά με τις προθέσεις ή και τις προσφορές των δύο αυτών χωρών της Κίνας και της Ρωσίας ως προς την δική σας πολύ όμορφη χώρα. Ευχαριστούμε. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής όπως και της ΕΕΔ. Η Επιτροπή. Όχι. Μάλιστα. Τότε θα επιστρέψω το μικρόφωνο στον κύριο Πρωθυπουργό. Παρακαλώ. Α, ζητώ συγγνώμη, δεν σας είδα εκεί πάνω. Δεν σας είδα. Ακόμα ένα μέλος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχα ζητήσει το λόγο και μετά είχα αλλάξει προς στιγμή γνώμη γιατί δεν μπορούσα να παραμείνω περισσότερο στην συνεδρίαση για λόγους άλλων δεσμεύσεων. Αλλά ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να θέσω μια ε, ερώτηση στον κύριο Πρωθυπουργό, ακόμα και δεν ακούσω την απαντήσή του. Παρουσιάσατε τον κατάλογο αυτών των προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη της χώρας, για το μέλλον της χώρας σας. Και καθορίσατε πόσο σημαντική είναι για εσάς η ειρήνη, η διαφάνεια, η καλή διακυβέρνηση, η ελευθερία και σε ποιο σημείο ε, είναι σημαντικό για σας να υπάρχουν, να οικοδομηθούν μάλλον και κάποιες ε, θεσμικές δυνατότητες όπως όλα αυτά. Εγώ ως συμπρόεδρος ε, της κοινοβουλευτικής συνδιάσκεψης με τις χώρες της Αφρικής και του Ειρηνικού και της Καραβικής θα, πρέπει να, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε σε διάφορες εταιρικέ σχέσεις και πλαίσια μαζί σας. Κύριε Πρωθυπουργέ, μιλήσατε για στρατηγική εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χώρα σας. Μια περιφερειακή εταιρική σχέση στρατηγική δεν θα ήταν πολύ πιο σημαντική για τη χώρα σας γιατί θα, θα σας επέτρεπε ίσως να οικοδομήσετε, να ενδυναμώσετε ακόμα περισσότερο την, την ειρήνευση και τις σχέσεις σας με τους γείτονές σας. Στο πλαίσιο που πολύ καλά περιγράψατε, Πρωθυπουργέ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον ε, κύριο Πρωθυπουργό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους αξιότιμους ε, βουλευτές για τις ερωτήσεις που έθεσαν. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση σχετικά με τον Νταρφούρ και την ε, μετεγκατάσταση των ε, εσωτερικά εκτοπιστέντων, τι είδου μέτρα λαμβάνουμε για να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη και γενικά πώς το βλέπουμε το όλο θέμα. Αυτή ήταν η ερώτηση. Κοιτάξτε, όσον αφορά την προσέγγισή μας στην, για την ειρνευτική διαδικασία, έχουμε συστήσει τέσσερις επιτροπές ή αν θέλετε τέσσερις ε, θεματικές ενότητες, ας τις πούμε έτσι, η μία αφορά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η δεύτερη ενότητα αφορά θέματα νομικής φύσεως, αποζημιώσεων και ε, δικαιοσύνης. Τρίτη ενότητα, πολιτικά θέματα, διακυβέρνηση και η τέταρτη ενότητα αφορά την ασφάλεια. Ε, βασική μας πρόθεση είναι να εξετάσουμε τα αίτια της σύγκρουσης ε, για να μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να θέσουμε τα θεμέλια για μια βιώσιμη ειρήνη. Οι εσωτερικά εκτοπιστέντες, οι πρόσφυγες, Αυτά είναι συμπτώματα μιας βαθύτερης κρίσης που εξανάγκασε τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους. Άρα δηλαδή πρέπει να ζητήσουμε τα βασικά αίτια αυτής της κρίσης και το προηγούμενο καθεστώς και οι εθνευτικές διαδικασίες ήταν σποραδικές, οι άνθρωποι συναντιόντουσαν κάπου σε κάποιες πρωτεύουσες, όμως ε, ε, τα συμφέροντα των πολιτών δεν λαμβάνονταν υπόψη. Αυτή τη φορά δεν πρόκειται να γίνονται μόνο επισκέψεις, αλλά ε, θα παρακολουθήσουμε τα συμφέροντά τους. Ε, θα διαβουλευτούμε με τους πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν πριν αρχίσουμε ε, τις διαπραγματεύσεις ξεκινήσαμε επισκέψεις επιτόπου. Είναι μακρύς ο δρόμος για να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη και μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω ότι η υποδοχή που μας επιφύλαξαν στις επιτόπιες επισκέψεις μας είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Επανήλθα, γύρισα στο Χαρτούμ με την εντύπωση ότι πραγματικά έχει προκύψει δυναμισμός, μια νέα κίνηση και θα το συνεχίσουμε αυτό. Δεν θα υπάρχει ειρήνη αν δεν μπορούμε να συνοηθούμε με τους πολίτες και θα το επιδιώξουμε. Το θέμα των σχέσεων με τον Νότιο Σουδάν, το πετρέλαιο και όλα τα σύναφη, το πετρέλαιο εξάγεται μέσα από τους αγωγούς και μέσα από το Βόρειο Σουδάν και το λιμάνι του Σουδάν και ελπίζουμε αυτό να, η διέλευση ε, και τα σημεία διέλευση γιατί είναι έξι περίπου τα σημεία διέλευση, ε, να μην αφορούν μόνο το πετρέλαιο, αλλά και τη διάβαση πεζών. Ήδη τρία έχουν ανοίξει τέτοια σημεία διέλευση. Οι εμπορικέ ανταλλαγέ μπορούν να βοηθήσουν και τι δύο πλευρέ, Αυτή τη γνώμη έχουμε ε, και ε, ε, μιλάμε για μια ζώνη ανάμεσα στις δύο χώρες. Όταν πήγα στο Νότιο Σουδάν και μίλησα με την ηγεσία της χώρας, συμφωνήσαμε ότι ε, αυτή ήταν μια κοινή μας επιθυμία, ότι θα πρέπει να μετατρέψουμε αυτά τα σύνορα σε σύνορα ειρήνης, ε, ευημερίας, ανάπτυξης, αντί να είναι τα σύνορα των συγκρούσεων. Ε, γιατί πολλά από αυτά τα σύνορα ε, δεν θα αλλάξουν ποτέ. Μπορούμε όμως να τα μετατρέψουμε σε ήπια σύνορα και να επιτρέπουμε τη διέλευση ανθρώπων και στις δύο πλευρές και δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Τώρα, για το θέμα των, ε, της φορολογίας και των δασμών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Σήμερα ε, έχουμε ένα 6% οι φόροι που είναι το εισόδημα από φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αλλά αυτό είναι απαράδεικτο. Ε, δεν μπορεί να επιβιώσει κανένα κράτος με αυτό το ποσοστό. Έχουμε τεράστια φοροδιαφυγή. Πάρα πολλές εταιρείε και που σχετίζονται με το δημόσιο δεν πληρώνουν καν φόρους. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε μια πολύ σημαντική μεταβατική και μεταρρυθμιστική διαδικασία. Ο Υπουργό Οικονομικών έχει συστήσει μια επιτροπή για φορολογική μεταρρύθμιση και αυτή την εβδομάδα θα συζητήσουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα και συστάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα της φοροδιαφυγής και θα προχωρήσουμε, θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τα αποτελέσματα που θα εξάγουμε. Ε, τόσα όσον αφορά την, ε, τα νερά του Νείλου, πώς μπορούμε να τα μοιραστούμε, το σχετικό φράγμα. Ε, είμαστε πολύ αισιόδοξοι σχετικά με αυτό. Το φράγμα ε, προσφέρει ευκαιρία και για το Σουδάν και για την Αίγυπτο να προχωρήσουν. Τρεις χώρες μπορούν να υποφεληθούν από το φράγμα και φαντάζομαι θα έχετε παρακολουθήσει τις ε, διαπραγματεύσεις ε, που έλαβαν χώρα την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον ε, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί καθορίσαμε ένα χάρτη πορείας μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, μία διαδικασία που θα μας επιτρέπει να συμφωνήσουμε για το θέμα του φράγματος το θέμα του χρονοδιαγράμματος και τις ρυθμίσεις γενικότερα για το φράγμα. Νομίζω ότι υπάρχει αποφασιστικότητα από πλευράς όλων για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το φράγμα. Τώρα, ε, την ερώτηση του ε, κυρίου από τη Βουλγαρία, ο ε, άνθρωπος τον οποίο αναφερθήκατε είναι και δικός μου φίλος και έχετε απόλυτα δίκιο. οι άνθρωποι που κατέβηκαν κατά χιλιάδες, κατά ε, εκατομμύρια στους δρόμους. Ναι, πράγματι έχουν ζήσει στερημένα, υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, αλλά το σύνθημα που ανέφερα προηγουμένως, το πρώτο του κομμάτι αφορά την ειρήνη. Ειρήνη, δικαιοσύνη και ε, ελευθερία. Ελευθερία, δημοκρατία, αυτά είναι λέξεις ε, κλειδί για αυτή την ε, περιοχή. Το Σουδάν ήδη από την αρχή, από τις αρχές της, από την αρχή της ανεξαρτησίας του, εδώ υπάρχει κάτι που δράτω με τις ευκαιρίες ε, για να το διορθώσω. Όταν μιλάμε για την Αφρική, λέμε ότι η Γκάνα ήταν η πρώτη ανεξάρτητη αφρικανική χώρα. Δεν είναι αλήθεια. Το 57 έγινε ανεξάρτητη Γκάνα. Το Σουδάν το 56, ένα χρόνο νωρίτερα. Δεν ξέρω. Ίσως ε, κάποιοι να μιλάνε γενικότερα για την υποσαχάρια Αφρική. Ε, το Σουδάν βρίσκεται στο βόρειο κομμάτι της υποσαχάριας Αφρικής. Τέλος πάνω. αυτό ίσως να είναι και δευτερεύον. Όμως το Σουδάν είναι μια παλόμενη ε, κοινωνία και κάθε φορά που αποκαθιστούμε τη δημοκρατία, τα πολιτικά κόμματα κινητοποιούνται, υπάρχουν πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Όπως σας είπα και προηγουμένως, ε, ηγούνται νέοι, πολλοί άνθρωποι και γι' αυτό το λόγο παραμένει ζωντανή η αλλαγή. Φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η δημοκρατία είναι μια αέναη διαδικασία. Ε, δεν μπορεί κανείς να τη μάθει. Πρέπει να την ασκεί. Δεν είναι, υπάρχει δηλαδή ένα μοντέλο που λέει αυτό είναι δημοκρατία και πάρτο και εφάρμοσέ το. Νομίζω αυτό που έχει σημασία είναι να την ασκεί κανεί στην καθημερινότητα με όλα τα δυσάρεστα συνεπακόλουθα. Ε, θεωρώ όμω ότι είμαστε αποφασισμένοι να συστήσουμε δημοκρατικού θεσμού. Ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Ε, Όπω σα είπα, αυτό δεν είναι μια γραμμική διαδικασία, αλλά θεωρώ ότι αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων που κατέβηκαν στου δρόμου ε, κινητοποιήθηκαν από αυτή την επιθυμία να συστήσουν μια δίκαιη χώρα με δημοκρατία, με σωστή διακυβέρνηση και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Τώρα, η άλλη ερώτηση που ετέθη. Μισό λεπτό σχετικά με την εκπαίδευση των νέων κοριτσιών, τις ευκαιρίες που έχουν. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πράγματι, αυτή είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όπως σας είπα, ξεκινάμε στο σωστό δρόμο. Θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίω δεν είμαστε ακόμα απόλυτα ικανοποιημένοι. Υπολείπονται ακόμα πολλά. Πρέπει να γίνουν πολλά. Κυρίως οφείλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε θέματα παιδείας, υγείας, αλλά κυρίως ε, σε θέματα εκπαίδευσης ε, των ε, νεαρών κοριτσιών, γιατί μόνο έτσι μπορεί να κερδίσει το κράτος. Και δεν έχουμε αυτά αυταπάτες. Προφανώς και υπολείπονται πάρα πολλά. Αυτό που είπατε στο τέλος που ρωτήσετε ε, πώς μπορεί να μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τη συνεργασία. Βοηθήστε μας, ε, χορηγώντας και εκταμιεύοντας κονδύλια για την εκπαίδευση, για την υγεία. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όταν μιλάμε για ιεράρχηση θεμάτων, το προηγούμενο καθεστώς, το 80% των κονδυλίων το διοχέτευε στον τομέα της ασφάλειας. Εμείς θέλουμε να το ανατρέψουμε αυτό. Επιθυμούμε οι επενδύσεις να γίνονται στην υγεία και την παιδεία. Και αυτό σημαίνει ότι θα αντιμετωπιστούν και θέματα που αφορούν στη διάκριση εις βάρος των γυναικών και πολλά σύναφη. Σχετικά με τη σχέση, γιατί ρωτήσατε, σχέση με την Κίνα και τη Ρωσία. Θέλω να πω ότι τις τελευταίες δεκαετίες η Κίνα ήταν ένας πολύ σημαντικός εταίρος του, του Σουδάν. Η Κίνα είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτη ε, στην ε, εκμετάλλευση του πετρελαίου, των κοιτασμάτων πετρελαίου στη χώρα μας. Ένα βασικό θέμα με την Κίνα είναι ότι το Σουδάν έχει ένα χρέος ε, περίπου 56 δις και ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού του χρέους αφορά την Κίνα. Αλλά η Κίνα εμπλέκεται και σε πάρα πολλά άλλα προγράμματα που υλοποιούνται στη χώρα. Είπα προηγουμένως ε, στις παρατηρήσεις που έκανα ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζουμε μια εξωτερική πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη της κατά κύριο λόγο τα συμφέροντα του Σουδάν. δεν θα φοβηθούμε να θέσουμε επιτάπητος ε, οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει έναντι οποιασδήποτε χώρα. Αυτό το χρωστάμε στους κατοίκους του Σουδάν. Ε, θέλουμε οι πολίτες ε, να είναι ένα κομμάτι του μέλλοντος της χώρας και θέλουμε επίσης, ε, πρώτα απ' όλα, όπως σας είπα, να ε, υπηρετήσουμε τα δικά μας τα συμφέροντα. Αυτό ε, είναι η αρχή που θα καθορίσει τη σχέση μας με την Κίνα και τη Ρωσία. Η τελευταία ερώτηση που τέθη, νομίζω από αυτού θέλω να πω το εξής οι συνεργασίες στην ευρύτερη περιοχή. Έχετε απόλυτα δίκιο οφείλουμε να διευθετήσουμε τα θέματα στην ε, περιοχή μας. Ίσως κατά παρελθόν να δημιουργήσαμε ε, προβλήματα σε όλους τους ε, γείτονες. Τώρα εγκαταλείπουμε αυτή την πρακτική, δημιουργούμε μία σχέση που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό. Και νομίζω με αυτή την αποφασιστικότητα θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες σχέσεις που θα μας ε, επιτρέψουν να υψώσουμε την φωνή της ε, λογικής, της ειρήνης και αυτό πράγματι ε, πρέπει να ξεκινήσει με τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με άλλες χώρες. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία για να συνεργαστούμε με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ε, και θα έχουμε ε, μια συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο πλαίσιο που υπάρχει, αλλά και πέρα από αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και να δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τέλος που μου δίνει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστούμε εξ ονόματο και των δύο επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που παραβρεθήκατε μαζί μα και που μα δώσατε πληροφορίε για την κατάσταση όσο έχει σήμερα στο Σουδάν. Μα ενημερώσατε για τι προτεραιότητέ σα και για τα σχέδιά σα, για το πώ θα μεταρρυθμίσετε και θα μεταμορφώσετε τη χώρα σα για να βρείτε δημοκρατικέ λύσει. Ω εκπρόσωπο χριστιανική χώρα στην Ευρώπη, Χαίρομαι επίσης που οι κόπτες, η κοπτική κοινότητα είναι κάτι που λαμβάνετε υπόψη στη χώρα σας, οι αρχές σας. Ελπίζω αυτό να αποτελέσει έναρξη των συνεργασιών μας που θα είναι, ελπίζω, επωφελής και για τη Σουδανική πλευρά αλλά και για την Ευρωπαϊκή πλευρά. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήλθατε εδώ στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ και έτσι λοιπόν λύεται τη σημερινή συνεδρία. Σας ευχαριστώ.